Είναι ο Γιάννου Βοζιβκέσκι ε, και οι δύο λοιπόν αυτοί οι βουλευτέ ορίστηκαν, διορίστηκαν στο ελεκτικό συνέδριο και τους ε, συγχαίρω